εξετάσετε να προταχθούν οι ομιλίες του ενός λεπτού για να μπορούμε να συμμετέχουμε πιο πολυπληθεί σε αυτές τις συζητήσεις όπως κάναμε και νωρίτερα. Καταγράφουμε αυτό το οποίο λέτε. Ξέρω ότι θα γίνει και μια συζήτηση για το θέμα αυτό και θα ληφθούν οι αρμόδιες αποφάσεις από την συζήτηση αυτή που πρέπει να γίνει μεταξύ των πρόεδρων των πολιτικών ομάδων. Πρώτο σημείο λοιπόν τώρα στην ημερήσια διάταξη είναι η δήλωση του Προέδρου σε σχέση με την αναγνώριση της γενοκτονίας στο Ρωμά κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ε, μέλη του Κοινοβουλίου, προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, η Ρωμά είναι πλέον η μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και η πιο καταπιεσμένη μειονότητα και αυτό ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου έτυχαν καταδίωξεις για φιλετικούς λόγους όπως και οι Εβραίοι. Και εκατομμύρια από αυτούς εξοντώθηκαν. Ήτανε πολίτες των ευρωπαϊκών χωρών για γενιές. Η 66η επέτειος της ε, απελευθέρωσης του Auschwitz-Birkenhof ήταν στις 22, 22 Φεβρουαρίου εφέτος και η Ρωμά ήταν η μεγαλύτερη ομάδα θυμάτων σε αυτά τα στατόπεδα. Δυστυχώ κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό ευρύτερα στου Ευρωπαίου. Μόνο μερικά κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αναγνωρίσει την εξόντωση των Ρωμά ω μορφή γενοκτονία. Είναι καιρό λοιπόν να αναγνωρίσουμε το γεγονό ότι οι Ρωμά πέρασαν από μια τραυματική εμπειρία γενοκτονίας και η παιδεία είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε την διάκριση εναντίον τους όπως και η ιστορική μνήμη. Πρέπει εμείς να αγωνιστούμε για τα δικαιώματα όλων αυτών των λαών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς σήμερα ενθυμούμεθα τους αδελφούς μας και τις αδελφές μας Ρωμά. Πρέπει όλοι να θυμηθούν τα βάσανά τους και να αγωνιστούν για μια καλύτερη κατανόηση της κατάστασής τους. It Ακολουθεί σύντομη συζήτηση. Σας παρακαλώ να μην αποχωρήσετε. Θα ακούσουμε το Συμβούλιο. Και ξέρετε ότι για την Ουγγρική Προεδρία το θέμα της ενσωμάτωσης στο Ρωμά είναι μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητές της. Θα ακολουθήσει η ομιλία του Αντιπρόεδρου της Κομισιόν και θα λάβουν το λόγο εν διαβραχαίων εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επίτροποι, Επίτροπε, ε, κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι βουλευτές, επιτρέψτε μου παρακαλώ να ξεκινήσω αναφέροντας ε, κάτι που είχε, πει, που είχε γράψει η Φρεντερικά Κόλομπαρ. Βρήκαμε τον πατέρα μου όταν φύγαμε από το Auschwitz στις 2 ε, Αυγούστου του 1945. Το όνομά του ήταν ε, ε, σε μια τεράστια λίστα ονομάτων. Δεν ξέραμε πού είχαν καταλήξει αυτοί οι άνθρωποι. Πολλοί κόσμος ε, μιλούσε για τον κίνδυνο μόλις, αλλά εμένα δεν με ένιωσαν οι κίνδυνοι αυτοί. Γιατί δεν είχα ε, την αίσθηση ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Θα ήθελα εξ ονόματος της Ουγγρικής Προεδρίας να συμφωνήσω με την ευγενή αυτή πρωτοβουλία η οποία αποσκοπεί να αποτίσουμε ε, φόρο τιμή στα θύματα του ολοκαυτώματος. Γιατί πρέπει να θυμούμαστε, γιατί δεν θέλουμε να ασχολούμαστε μόνο με το μέλλον. Ένας Αμερικανός ε, ε, ιστορικός, ο Τζορτ Σανταϊάννα, είπε ότι όποιος δεν είναι σε θέση να θυμάται το παρελθόν, είναι καταδικασμένος να επαναλαμβάνει το παρελθόν. 220.000 ε, Ρώμα και Σύντι ήταν οι πιο μετριοπαθείς ε, αν θέλετε εκτιμήσεις ε, για τα άτομα που δολοφονήθηκαν. Μιλάμε για Ούγγρους, Γερμανούς, Γάλλους, Πολωνούς, Σέρβους, πολίτες. Πολλοί οι άντρες, πολλές γυναίκες, πολλά παιδιά, οι οποίοι αν θα ακόμα σήμερα, θα ήταν Ευρωπαίοι πολίτες. Οι επιζήσαντες αναφέρουν ότι στο Auschwitz ε, επέτρεπαν στους ε, Ρωμά να ζουν μαζί. Δεν τους χώριζαν. Μέχρι τις 2 Αυγούστου του 1944, εκείνη τη νύχτα, 2.000 ε, φυλακισμένοι δολοφονήθηκαν, εκτελέστηκαν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξαναγεννήθηκε μετά τον εφιάλτη της ΣΟΑ και του Ποραγιάμος. Το ευρωπαϊκό όραμα συνενώνει τους λαούς της Ευρώπης για να αποκηρύξουν αυτά που έγιναν το, στο Auschwitz. Και αυτό αποτελεί ακόμα τμήμα του παρελθόντος. Θα αναρωτηθεί κανένας πιο είναι το μέλλον. Η Ουγγρική Προεδρία θεωρεί ότι θα πρέπει να συζητάμε μαζί και το παρελθόν και το μέλλον. Ο Βίκτορ Όρμπαν παρουσίασε αρχές Ιανουαρίου το πρόγραμμα της Ουγγρικής Προεδρίας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δήλωσε ότι η στρατηγική για τους Ρωμά αποτελεί προτεραιότητα της Ουγγρικής Προεδρίας. Γιατί η Ευρώπη μπορεί να είναι έξυπνη και ευφύης, αλλά να μην έχει καρδιά. Καρδιά θα έχει μόνο αν φροντίσει και πραγματοποιήσει τελικά την κοινωνική ενσωμάτωση, ενοποίηση. Εγώ θα ήμουν προσωπικά πολύ υπερήφανη αν όλοι στο τέλος της ε, Ουγγρικής Προεδρίας μπορούμε να μιλούμε για μια κοινή στρατηγική για τους Ρωμά. Και ευχαριστούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει. Το Συμβούλιο και η Ουγγρική Προεδρία θέλουν να συνδράμουν και αυτοί. Θέλουμε να συμβάλλουμε προκειμένου όλοι να θεωρούν ότι η Ρωμά, ακριβώς όπως και όλοι οι άλλοι λαοί του κόσμου, δεν, είναι, δεν αποτελούν πρόβλημα, αλλά αποτελούν μια χρήσιμη πολιτισμική οικονομική ε, πηγή. Thank you, Madam Minister. Ε, Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Έχει το λόγο ο Μάρος Σεφκοβίτς, ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν τώρα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πριν από λίγες μέρες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, εόρτασε την ημέρα ενθύμησης του ολοκαυτώματος μαζί με τους επιζήσαντες αυτής της τραγωδίας. Και είναι πρέπον σήμερα να θυμηθούμε την γενοκτονία των Ρωμά μετά από το Yad Vashem, μετά από το Μουσείο του Ολοκαυτώματος στο, στο, στη Washington στην Αμερική, βλέπει κανείς πραγματικά πόσο ικτρή ήταν αυτή η καταστροφή το Ρωμά. Αυτή που έχετε δει το μνημείο στην Ιερουσαλήμ, νιώθετε πραγματικά κλονισμό και καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατο μόνο πριν από 70 χρόνια να είχε γίνει κάτι τέτοιο στην Ευρώπη. Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει να συζητήσουμε για τα θέματα αυτά. Πρέπει μάθουν τα παιδιά μας για αυτή την τραγική ιστορία της Ευρώπης, γιατί η ιστορία έχει την τάση να επαναλαμβάνεται. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να εξασφαλίσουμε απόλυτα ότι αυτή η τραγωδία θα μείνει στη μνήμη των ανθρώπων για να μην επαναληφθεί. Θα πρέπει να αγωνιστούμε όλοι για να ξεπεράσουμε τα φαντάσματα του παρελθόντος. Η ιστορία μας έχει δείξει ένα μεγάλο μάθημα για το τι μπορεί να κάνει το μίσος και η μυσαλλοδοξία. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση εδράζεται σε θεμελιώδη δικαιώματα και αξίες που περιλαμβάνουν την προστασία των μειονοτήτων, την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας και την απαγόρευση των διακρίσεων. Όλα αυτά εφαρμόζονται πλήρως στους Ρωμά. Είναι απαράδεκτο στον 21ο αιώνα οι Ρώμα να πρέπει ακόμα να αντιμετωπίσουν διακρίσει επί τη βάση τη εθνοτική του προέλευση. Είναι πάρα πολλοί Ρωμά ακόμα που αντιμετωπίζουν ρατσισμό, διακρίσει και κοινωνικό αποκλεισμό. Πάρα πολλά παιδιά των Ρωμά είναι στου δρόμου και όχι στο σχολείο. Πάρα πολλοί Ρώμα δεν έχουν ακόμα πραγματικέ ευκαιρίε να εργαστούν και πάρα πολλέ γυναίκε Ρωμά είναι θύματα βία και εκμετάλλευση. Η συμπέριληψη στο Ρωμά είναι προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και απαιτεί την δέσμευση και την κοινή δράση τοπικών και εθνικών αρχών τη κοινωνία των πολιτών και των θεσμών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη δική τη πλευρά, η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι απόλυτα προσιλωμένη στην επίτευξη τη ενσωμάτωση των Ρωμά στι κοινωνίε μα. Εργαζόμαστε προ αυτή την κατεύθυνση εδώ και πολύ καιρό και αυτό είναι μια μακροπνοή στρατηγική για μα. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι κατά κύριο λόγο η ευθύνη της ενσωμάτωσης στο Ρωμά βρίσκεται στα χέρια των κρατών μελών. Γι' αυτό τους έχουμε δώσει ένα συγκεκριμένο κατάλογο δράσεων που θα μπορέσουν να κάνουν πιο αποτελεσματική τη δράση τους υπέρ των Ρωμά στην ανακοίνωση Κομισιόν πέρσι που ήταν το πρώτο έγγραφο πολιτικής που αφορούσε ιδιαίτερα αυτή τη μειονότητα. Η αξιολόγησή μας όμως δείχνει ότι τα κράτη-μέλη χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των πολιτικών τους για την ενσωμάτωση των Ρωμά. Γι' αυτό η Κομισιόν <clears throat> μαζί με την Ουγγρική Προεδρία θα εγκρίνει τον Απρίλιο ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις εθνικές στρατηγικές ενσωμάτωσης των Ρωμά και θα κάνει προτάσεις έτσι για να αντιμετωπιστεί ο αποκλεισμό τους από τις κοινωνίες. Για να κλείσω αυτήν την επίσημη στιγμή θα ήθελα να τονίσω από την πλευρά της Κομισιόν την ανάγκη να υποστηρίξουμε τα, και να προστατέψουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών και να εξασφαλίσουμε την αρμονική ενσωμάτωση όλων των πολιτών στην κοινωνία μας. Είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι η ιστορία δεν θα επαναληφθεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, τώρα εξ του ΕΛΚ, η κυρία Λίβια και Γιαρόκα. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι. Εξ ονόματος του ΕΛΚ θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίηση και ευγνωμοσύνη μου για το γεγονός ότι για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μιλάει για τη μνήμη της θυσίας των Ρωμά. Νομίζω ότι ήταν, είναι καθήκον μας να θυμόμαστε το παρελθόν και να παίρνουμε διδάγματα από αυτό. Όσο δύσκολα και να είναι τα μαθήματα που πρέπει να πάρουμε και αυτά τα μαθήματα πρέπει να τα διατηρούμε στη συλλογική μας μνήμη. Ξέρω ότι πολλά ιδρύματα, ερευνητικά ιδρύματα συμβάλλουν στην διερεύνηση του τι ακριβώς έγινε στο παρελθόν και την καταγραφή. Σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα πρέπει να βλέπουμε όλους τους αιώνες πόσους αιώνες μάλλον ιστορίας μοιραζόμαστε με τους τσιγκάνους και γι' αυτό πρέπει πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή να τις ενθαρρύνουμε. Σήμερα η Ρωμά είναι ελεύθεροι πολίτες ισότιμοι με τους υπόλοιπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωστό και δίκαιο. Έχουμε τουλάχιστον 7 αιώνες κοινή ιστορίας και οι Τιγκάνοι έχουν υπάρξει πιστοί στην κάθε τους πατρίδα παρά τον αποκλεισμό και το μίσος που έζησαν καθόλου στους αιώνες αυτούς. Πρέπει λοιπόν να μπορέσουν να ζήσουν σε ειρηνική συνύπαρξη με όλους τους υπόλοιπους. Γνωρίζουμε λοιπόν το παρελθόν και ελπίζουμε να υπάρξει αυτή η συμβίωση γιατί μόνο με αυτό μπορεί να επιβιώσει η κοινότητά τους και οι υπόλοιπες μαζί ώστε ο κόσμος να γίνει καλύτερος. Οι χώρες μας κατάφεραν να συμβιώσουν και να συνεργαστούν και σε θέματα πολύ σοβαρά και αυτό θα ήθελα να προσθέσω μόνο το εξής. Σε δύο εβδομάδες θα εξετάσουμε το θέμα μιας στρατηγικής για τους Ρωμά και ελπίζουμε και αυτό κάποτε να επιτυχθεί. Ευχαριστώ πολύ, ο πρόεδρο. Τώρα, εξ τη Σοσιαλιστικής και δημοκρατική Ομάδας, ο Αντιπρόεδρος της Ομάδας αυτής, κ. Χάνε Φόβοντα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας ε, ευχαριστώ και εσάς και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και τον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν για τη θέση που έλαβαν για το θέμα αυτό. Η στιγμή αυτή είναι πολύ σημαντική. Εξ όμως της ομάδας μου θα λάβει το λόγο και η Κίνγκα Γκάλ. Η σφαγή, η γεροκτονία των Ρωμά είχε κάπως τεθεί στο περιθώριο σε σχέση με την εξόντωση των Εβραίων. Αλλά είναι και αυτοί όπως και οι Εβραίοι θύματα του ε, ναζιστικού καθεστώτος και φυσικά και οι ομοφιλόφιλοι είναι και αυτοί θύματα τα οποία εξοντώθηκαν κατά τη διάρκεια της ναζιστικής εποχής. Συμφωνώ με την Ουγγρική Προεδρία ότι η καλύτερη μορφή ανάμνησης είναι να σκεφτόμαστε όχι το παρελθόν μόνο, αλλά και το μέλλον. Η κατάσταση των Ρωμά στην Ευρώπη δεν είναι ικανοποιητική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι θύματα πάντα διακρίσεων, είναι θύματα προκαταλήψεων. Υπάρχει μια χώρα η οποία θεωρεί ότι πρέπει να αλλάξει το όνομά του και αντί για Ρωμά να του λέει Τσιγκάνου. Δεν το λέω αυτό για να επικρίνω. Απλώς για να δείξω την ανάγκη που πρέπει που υπάρχει για να αντιμετωπίσουμε την διάκριση και την ε, προκατάληψη και όχι να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε ονόματα σε αυτές τις μορφές διακρίσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τις επισκέψεις που κάναμε και σε πολλές ε, χώρες είδαμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με τους Ρώμα. Υπάρχει ένας φαύλος κύκλος διάκρισης, θέση σε μειονεκτική θέση που δεν σπάει ποτέ. Πάρα πολλά παιδιά πηγαίνουν ακόμα σε χωριστά σχολεία των Ρωμά. Και χαίρομαι πάρα πολύ για το γεγονός ότι η Ουγγρική Προεδρία έθιξε και αυτό το θέμα. Και παρά τις διαφορές που μπορεί να έχουμε μαζί σας, κυρία ε, Πρόεδρε της ε, Ουγγρικής, κυρία, ε, Ουγγρικής Προεδρίας, θα σας υποστηρίξουμε απόλυτα για τα θέματα αυτά. Ξέρετε ότι ο Γκίντερ Γκράσ, ο μεγάλος γερμανός συγγραφέας, έχει ιδρύσει και ένα ίδρυμα για τους Ρώμα που τονίζει ότι αυτοί λόγω της διασποράς τους, λόγω της μετακίνησής τους είναι πραγματικοί Ευρωπαίοι γιατί έχουν περάσει όλη, όλη την έκταση της Ευρώπης και έχουν παίξει σημαντικό ρόλο και στην διαμόρφωση της οικονομίας τους η δραστηριότητά τους, το γεγονός ότι περάσαν τα σύνορα τόσο συχνά στην Ευρώπη έχουν βοηθήσει να δημιουργηθεί και το ευρωπαϊκό ε, αυτό πνεύμα και θα πρέπει τα δικαιώματά τους από την Πορτογαλία ως τη Ρουμανία να τύχουν εγγύησης. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να νιώθουν στο σπίτι του οι Ρωμά, να έχουμε όλες τις προϋποθέσεις ώστε να μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα χωρίς να τους εμποδίζουν ή να τους στέλνουν πίσω. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ αυτό το οποίο έκαναν οι Ναζί, την φρικτή αυτή εξόντωση των Ρωμά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα η κυρία Ρενάτε Βέιμπερ εξ ονόματος της Άλντε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σαμενταρέμπεον ε, στα ρωμανικά ε, σημαίνει εφιάλτης επιγής και αυτό έζησαν οι Ευρωπαίοι Ρωμά κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου όταν εκατοντάδες χιλιάδες δολοφονήθηκαν πολύ απλά επειδή ανήκαν στην ε, εθνοτική κοινότητα των Ρωμά. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πόσοι ήταν στον αριθμό. Άλλοι λένε ότι ε, είναι 250.000 τα θύματα, άλλοι μιλούν για ένα εκατομμύριο θύματα. Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα επειδή δεν υπήρξε ε, σαφήνεια, δεν, υπήρξε, δεν ήταν σαφές πόσοι χάθηκαν στο ολοκαύτωμα των Ρωμά επί σειρά ετών αγνοούνταν συστηματικά τα άτομα αυτά και γι' αυτό το λόγο σήμερα η σημερινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την φωνή του Προέδρου αποτελεί μια ιστορική στιγμή. Δεν θα πρέπει όμως να περιοριστούμε σε αυτή τη στιγμή. Αυτή η στιγμή θα πρέπει να ακολουθηθεί από συγκεκριμένα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών. Είναι απαραίτητο η αναγνώριση αυτή της γενοκτονίας των Ρωμά γίνει από κάθε χώρα και θα πρέπει να προωθηθεί η επίγνωση της πτυχής αυτής της ιστορίας προκειμένου τα παιδιά της Ευρώπης να γνωρίσουν, να, μάθουν για το ολοκαύτωμα να μάθουν για τις ε, αιώνες που οι Ρωμά ήταν σκλάβοι. Όσο του η ευρωπαϊκή κοινωνία συνειδητοποιήσει ότι έχουμε αυτό το ιστορικό καθήκον προς την κοινότητα αυτή, δεν θα καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε το ρατσισμό, ούτε θα πετύχουμε με τις εθνικές και ευρωπαϊκές μας στρατηγικές για τη συμπερίληψη των Ρωμά και την ενσωμάτωση των Ρωμά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Γκρέζ από τους Πράσινους. Με βαθιά συγκίνηση λαμβάνω το λόγο σήμερα αυτό το απόγευμα ενώπιον τη Ολομέλη. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σα ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τη δέσμευσή σα. Η αναγνώριση τη γενοκτονία των Τσιγκάνων είναι μια ιστορική στιγμή για τα εκατομμύρια Ευρώπων των ανθρώπων που ταξιδεύουν, των Μανούς, των Σιντί, των Ρωμά. Χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων σκοτώθηκαν τα σκοτεινά χρόνια του νασισμού πολλές φορές με την ετικέτα, με τη ρετσινιά των ακοινωνικών ατόμων. Αυτό είναι η κοινή ιστορία όλων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να το θυμηθείτε ότι οι Τσιγκάνοι ήταν οι πρώτοι οι οποίοι από τη μία χώρα στην άλλη χώρα της Ευρώπης προτού να υπάρξει η ελεύθερη κυκλοφορία και ο κοινό χώρος της Ευρώπης. Σήμερα εκπροσωπούν ένα πληθυσμό περίπου 10 εκατομμυρίων ατόμων, είναι η πιο μεγάλη μας μειονότητα και η θλιβερή τους ιστορία είναι και θλιβερή ιστορία της Ευρώπης. Είναι καιρό, αγαπητοί, καιρός αγαπητοί συνάδελφοι να δώσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους σε αυτούς τους πολίτες. Εμπιστοσύνη και στον εαυτό τους αλλά και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο περιθώριο, που είναι καταδικασμένοι όχι μονάχα στην ιστορία του πολέμου αλλά και στην σιωπή και την άγνοια σε σχέση με την τύχη που είχαν στο Δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο. Η αναγνώριση της γενοκτονίας των Τσιγκάνων είναι μια πραγματικά μια πράξη μνήμης. Θα πρέπει να είναι και το δείγμα και η απόδειξη μια θέληση για ένα διαφορετικό μέλλον. Οι Ευρωπαίοι κοινοβουλευτικοί στην Ανατολική και στη Δυτική Ευρώπη την προηγούμενη εβδομάδα στην Bundestag έχουν αναλάβει τι ευθύνε του σε σχέση με την ιστορία με το να αποδεχθούν την αναγνώριση της γενοκτονίας. Είναι ένα πρώτο βήμα για να έχουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση των Ευρωπαίων πολιτών έναντι της μειονότητας των Ρωμά. Είναι μακρός ο δρόμος, αλλά θα πρέπει, μακρύς ο δρόμος, αλλά θα πρέπει να τους κάνουμε πλήρης πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρώμα. Ε, Σας ευχαριστώ. Μάρκ Μιγκάλσκι για την ομάδα των συντηρητικών. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Το γεγονός ότι οι Ρωμά υπήρξαν θύματα γενοκτονίας κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είναι προφανές όσο προφανές τουλάχιστον και αυτό που ισχύει για τους Εβραίους και όποιος το αρνείται θα πρέπει να θεωρείται ψεύτης όπως γίνεται και για όποιον αρνείται τη γενοκτονία των Εβραίων. Η Πολωνοί ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα των θυμάτων και θα έπρεπε να θυμηθούμε όλα τα θύματα του ολοκαυτώματος κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στο Auschwitz και στα υπόλοιπα στατόπεδα συγκέντρωσης θυμίζουν και τις δολοφο... μαζικές δολοφονίες στο Κατίν Όλα αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε και να εορτάζουμε τη μνήμη τους για να μην ξανασυμβούν ποτέ. Το κοινοβούλιο μας έχει την ηθική υποχρέωση να διασφαλίζει ότι θα τα θυμόμαστε όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για όσα είπατε. Η Κορνηλία Έρνστ εξ ονόματος της ΓΚΟΕ. Κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ώρα σήμερα και πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, αποτείγουμε φόρο τιμή στο ολοκαύτωμα το Ρωμά και το Συντινά. Ας σα αναφέρω κάτι, ε, ένα αποχαιρετιστήριο γράμμα το οποιο ένα ένας 14χρονο ε, απέστειλε το 1944 στο Auschwitz και έγραψε ότι ξαναβρήκα του γονεί μου. Βρισκόμαστε στο στρατόπεδο συγκέντρωση. Σας ευχαριστώ για όλα όσα μου για όλα όσα κάνετε για μένα και τα ξαναλέμε στους ουρανούς. 5.000 Ρώμα και Σύντη δεν ξαναγύρισαν στα σπίτια τους και παρά το γεγονός ότι ήταν τα πρώτα θύματα η Ρώμα και η Σύντη, σήμερα 66 χρόνια αργότερα δεν έχει υποθεί ακόμα ξεκάθαρα η πλήρης αλήθεια και το πόσο ε, συμμετείχε και η όλη κοινωνία. Χρειαζόμαστε μια σαφήνεια για αυτό το θλιβερό κεφάλαιο της ιστορίας. Θα πρέπει να το χαρακτηρίσουμε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, προκειμένου να μην επαναληφθεί η ιστορία αυτή. Οι προκαταλήψεις κατά των ανθρώπων αυτών θα πρέπει να καταπολεμηθούν και οι φασιστικές ιδεολογίες, όπως για παράδειγμα πρόπερση στην Ουγγαρία, όπως εκδηλώθηκαν πρόπερση στην Ουγγαρία, θα πρέπει να καταπνιχτούν με το κουράγιο των πολιτών. Η αλληλεγγύη δεν αποτελεί ε, πλέον έκτημα για λίγους, αλλά δικαίωμα για όλους. Ε, pani Σαβέλα, Wolność i Demokracja. Θα ήθελα να ενώσω κι εγώ τη φωνή μου με αυτά τα οποία έχουν υποθεί μέχρι τώρα. Οι Ρωμά έχουν συνεισφέρει καθοριστικά και στην ανάπτυξη της Ευρώπης και ιδιαίτερα στον πολιτισμό της. Αυτό που θα ήθελα να παρατηρήσω ορθολογικά κύριε Πρόεδρε είναι ότι οποιαδήποτε προγράμματα αφορούν τους Ρωμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προέρχονται από την Επιτροπή έχουν έναν κατακαιρματισμό. Ε, συνήθως συμπεριλαμβάνονται ε, μέσα στον κοινωνικό αποκλεισμό. Η πρότασή μου θα ήταν για μια ορθολογική προσέγγιση για να πούμε ωραία τα λέμε ωραία εδώ αλλά τι κάνουμε κιόλας. Η πρότασή μου είναι η Κομισιόν να υιοθετήσει ένα initiative μόνο για τους Ρωμά, να το βγάλει από τον κοινωνικό αποκλεισμό και να είναι ένα project το οποίο αφορά και μόνο τους Ρωμά. Έτσι θα μπορέσουμε να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά σε εθνικό επίπεδο για τους Ρωμά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Uh, uh Ευχαριστώ. Αυτό είναι το τέλος της συζήτησής μας. Ευχαριστούμε την Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. Κύριε Αντιπρόεδρε της Κομισιόν, επίσης σας ευχαριστούμε και όλους τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους και τα σχόλιά τους αυτήν την τόσο σημαντική για όλους μας συζήτηση, σημαντική για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαν σύνολο. Κλείνουμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση. Το επόμενο σημείο της σημερινής διάταξη είναι η δηλώση του Συμβουλίου και της Κομισιόν για την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τη 4 η Φεβρουαρίου 2011.